Την ε, νομική επιτροπή που είναι αρμόδια για το θέμα. Επίσης έλαβα από τις ομάδες ΕΛΚ πολλά αιτήματα τροποποίηση στις ε, κοινοβουλευτικέ επιτροπές και τι διακοινοβουλευτικέ αντιπροσωπείες. Ο κατάλογος αυτών των ε, ονομάτων θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά της Συνόδου. Εάν ε, πριν από την έγκριση της ημερήσιας διάταξης δεν υπάρξουν παρατηρήσεις, οι διορισμοί αυτοί θα υιοθετηθούν. Η αρμόδια επιτροπή έχει παρουσιάσει μια διόρθωση σε σχέση με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αυτή οθετήθηκε σε δεύτερη ανάγνωση και αυτή θα δημοσιευθεί στα πρακτικά.